All on holidays. κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω την κύρια Αστόν, την υψηλή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και αντιπρόεδρος της Κομισιόν στη συνεδρίασή μας ως ε, ε, επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Θα μας παρουσιάσει τις συζητήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών αυτή τη εβδομάδα. Κύριε Άστον, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι ε, πολλές φορές έχετε, είχατε στο παρελθόν δυσκολία να είσαστε μαζί μας λόγω αντικρουμένων υποχρεώσεων, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επισκόπηση που θα κάνετε για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και θα υπάρχει δυνατότητα οι βουλευτές να σας θέσουν ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις. και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό για μας να γνωρίσουμε ποια είναι η κατάσταση χωρίς να σας ε, υπερφορτώσουμε ιδιαίτερα με τις ερωτήσεις μας. Ξέρουμε ότι το θέμα της Συρίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή. Όλα τα θέματα της ε, αντιπαράθεσης στην ε, Μέση Ανατολή, επίσης τα θέματα του Αφγανιστάν τα θέματα της γειτονία με τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης. Μας ενδιαφέρει σε όλα αυτά τα θέματα να δούμε ποια είναι η εξέλιξη και ιδίω οι εξέλιξεις οι πρόσφατες στη Συρία και στο Κωσυφοπαίδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για το γεγονός ότι έχετε προωθήσει αποφασιστικά τις επαφές με το... για το θέμα της Συρίας και του Κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο και ελπίζουμε το... ότι τώρα θα μπορέσουν να γίνουν ε, σύντομα αποφάσει στα θέματα αυτά και επίσης το θέμα της ε, υποψηφιότητας της Τουρκίας. Η παρέμβασή σας, η θέση σας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Θα έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με την Τουρκία, με το προσδοκόμενο άνοιγμα ενός κεφαλαίου, με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Όλα αυτά φυσικά εξαρτιόνται και από την εσωτερική πρόοδο στην Τουρκία και επίσης μπορείτε να αναφέρετε και για το πρόσφατο ταξίδι σας στην Αίγυπτο. Είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο ίσως θα μας απασχολήσει σε κάποια άλλη στιγμή πιο ε, εκτενώς, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε και το θέμα αυτό, ιδίω για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο. Είναι παρόν ο κύριος ε, ε εδώ, ο οποίος είναι ε, επικεφαλής μιας τέτοιας ΜΚΟ και επομένως έχουμε το πρόβλημα αυτό των ΜΚΟ οι οποίες βρίσκονται στην Αίγυπτο και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους. Και έχουμε πολλούς ε, από τις ε, ΜΚΟ αυτούς που ή απειλούνται ή βρέθηκαν ορισμένοι από αυτούς στην φυλακή. Και αυτό αφορά και το Ίδρυμα Κόναρντ εγώ ήμουν το Σάββατο στο Κάιρο. Είδαμε να υπάρχουν και διαδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Αίγυπτο και υπήρξαν πολλές υπογραφές οι οποίες συνελέγησαν εναντίον του Πρόεδρου Μόρση. Όλα αυτά φυσικά είναι αποφασιστικά γεγονότα για την περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων που έχουμε με την Αίγυπτο και την σταθερότητα στην περιοχή. Σας δίνω το λόγο κυρία Άστον. Well, uh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι ήταν μαζί σας η Χέλγκα Σμιτ που αναφέρθηκε στα του Ιράν μετά από την μη αναμενόμενη νίκη του Χασάν Ροχάμι. Θα ήθελα να συνεχίσω στην δική της ε, θα έλεγα γραμμή και όθηση. Ελπίζω ε, να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τον υπόλοιπο κόσμο ε, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων της διαδικασίας 3 3 προσπαθούμε να δούμε τι θα μεσολαβήσει μέχρι τις αρχές Αυγούστου που θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Θα ξεκινήσω από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις επίσης. Ε, θα ξεκινήσω με την Τουρκία. Γνωρίζω από τις συζητήσεις που είχαμε στην Ολομέλεια πριν λίγο καιρό πόσο ανησυχείτε για τα τεκτενόμενα στη χώρα αυτή πρόσφατα, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι αρχές καταστολής εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών. Είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και όσοι είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να υποστούν τις κυρώσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις επαφές με την Τουρκία ε, για να επηρεάσουμε ε, την κατάσταση, να λειτουργήσουμε σαν μοχλός και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ήδη έχουμε ε, πει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έτσι ώστε και οι φωνές, οι φωνές της αντιπολίτευσης και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν να εκφραστούν. Θα πρέπει οι σχέσεις μας με την Τουρκία να αναπτυχθούν στα πλαίσια μιας πορείας η οποία θα δίνει νέες δυνατότητες έτσι ώστε οι αξίες και ο τρόπος με τον οποίο εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και στον τομέα του κράτους δικαίου και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνουν κοινές. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων λοιπόν αποφάσισε να ανοίξει το κεφάλαιο 22 και όπως βλέπετε θα γίνει η διακυβερνητική μετά την παρουσίαση της εκθέσεως της ετησίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή λύση, κρατά αν θέλετε την διαδικασία αυτή και ταυτόχρονα επιτρέπει ε, να βελτιωθούν οι σχέσεις. Εμείς είδαμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τη συνάντηση κορυφής για την πολιτική γειτονία. Εμείς συζητήσαμε τα θέματα των σχέσεων με τους γείτονες, με τις γειτονικές χώρες. Είχαμε και μια συνάντηση μάλιστα των Υπουργών της Ανατολικής Γειτονίας, θα έχουμε μάλλον στις 17 Ιουλίου. Αυτό το κάνουμε για να δείξουμε τη σημασία που ε, δίδουμε στις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές, ε, να προετοιμάσουμε σωστά τη συνάντηση κορυφής και να ενθαρρύνουμε αν θέλετε και την ε, διαδικασία και την αίσθηση του ανήκειν σε αυτήν την ομάδα έτσι ώστε να διαχειριστούμε τις φιλοδοξίες που υπάρχουν. Το Συμβούλιο ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και το τι θα κάνουμε μετά τη συνάντηση του Βίλνιους, ποια θα είναι η στρατηγική μας και οι φιλοδοξίες μας για τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσει τη συνάντηση του Βίλνιους. Ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει σε εταιρικέ σχέσεις και συζητήσεις με τη Μολδαβία, την Αρμενία, την Ουκρανία. Δεν χρειάζεται να θυμίσω ότι η Ουκρανία παρουσιάζει ορισμένα θέματα στα οποία απαιτείται περαιτέρω πρόοδος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή στο Βιλνίους εφόσον η Ουκρανία σταθεί στα επίπεδα τα οποία έχουν ε, δοθεί από το Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Ανησυχούμε όμως για το κράτος δικαίου και για επιλεγμένα θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και θα θέλαμε να ξεκαθαριστούν ε, τα πράγματα αυτά λίγο. Παράλληλα συνεχίζουμε τη συζήτηση για την ε, σημασία που έχουν οι σχέσεις με τη Λευκορωσία και εννοούμε κυρίως την κοινωνία των πολιτών και το πόσο θα επηρεάσει το θέμα αυτό τις συζητήσεις που θα γίνουν στο ε, Βίλνιους. Συζητήσαμε και τα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών. Εγώ έκανα μία εισαγωγή σχετικά με αυτό που ονομάζουμε οριζόντια ή σφαιρικά θέματα. Έγιναν κάποιες συζητήσεις για την ενέργεια και αυτή είναι η δεύτερη συζήτηση για τις κλιματολογικές αλλαγές. Ζητήσαμε από την Αρμόδια Επίτροπο να είναι μαζί μας. Θέλουμε το θέμα αυτό να τίθεται συστηματικά στις συζητήσεις μας με τρίτες χώρες, όχι μόνο από τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ή από εμάς, αλλά και από όλους τους υπουργούς έχει σημασία κάποιοι κομβικοί εταίροι μας, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείες, ε, να θεωρήσουν ότι υπάρχει εδώ μια επίγουσα ανάγκη αντίδρασης έτσι ώστε να το εντάξουμε το θέμα αυτό στην γενική ε, εξωτερική πολιτική. Λόγω αυτών που συμβαίνουν ε, σε θέματα ε, κλιματολογικών αλλαγών υπάρχουν αρνητικές δραματικές συνέπειες για δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο και χώρες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν σε ε, συμβάντα φυσικά όπως το τσουνάμι, όπως οι πλημμύρες κτλ. Το 2015 θα γίνει μια μεγάλη συνέλευση στο Παρίσι και ζητήσαμε από την Επίτροπο να επανέλθει με μία πρόταση για το τι θα πρέπει να γίνει ε, ε, μέχρι τότε. Χρειαστήκαμε κάποιο χρόνο για να δούμε και τα θέματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή να προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιες κινήσεις και βελτιώσεις λόγω και της τεράστιας εξαιρετικής προσπάθειας την οποία έχει αναλάβει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κέρι. Εμένουμε στις λύσεις που είχαμε προκρίνει στο παρελθόν και υποστηρίζουμε τις τρέχουσες διαδικασίες. Είμαστε σε τακτική αν όχι μόνιμη επαφή με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τις υπηρεσίες του Υπουργού Κέρι και θέλουμε να στηρίξουμε πλήρως τις προσπάθειές του λέγοντας ότι αν ήταν εδώ θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει στις προσπάθειες αυτές και πολιτικά και οικονομικά όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι και είχα πάει στην Ιερουσαλήμ και την Ραμάλα την προηγούμενη εβδομάδα. Συναντήθηκα με την πολιτική ηγεσία, συναντήθηκα επίσης και με τον Νετανιάχο, πήγα στην... Πήγα στη Γάζα, μάλιστα ήταν η μέρα των προσφύγων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα των προσφύγων είναι ένα τεράστιο θέμα όχι μόνο σχετικά με την Συρία σήμερα, αλλά πολύ γενικότερα στον πλανήτη μας. Και ήταν ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούμε να βοηθάμε τα παιδιά, ας πούμε, στην Γάζα, στον τομέα της εκπαίδευσης και γενικότερα της οικονομίας. Αλλά αυτά θα επανέλθουν στη συζήτηση τον μήνα Ιούλιο, γιατί το Συμβούλιο σίγουρα θα θέλει να εξετάσει εκ νέου το θέμα μετά από βήματα προόδου ελπίζω που θα έχουν σημειωθεί από τον Υπουργό Κέρι. Ζητήσαμε να συναντηθούμε και στο γεύμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ράσμουσεν. Έχω τακτικές διμερείς συναντήσεις μαζί του και διοργανώνονται επίσης και τακτικές υπηρεσιακές συναντήσεις με την Γραμματεία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Το θέμα που συζητήσαμε μαζί του είναι το μέλλον του Αφγανιστάν. Μας υπενθύμησε τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών και της ασφάλειας. Μας τόνισε επίσης και τη σημασία που δίδει στην, στον έντονο χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η συνεργασία μας, τη συνεργασία τη στρατιωτική με τις αρχές του με, με τον Αφγανικό στρατό και τις ε, ε, αυγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Ε, Πέμεινε επίσης και στη μεγάλη σημασία που θα έχει η εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ μετά το 2014 στη χώρα του Αφγανιστάν και καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ΝΑΤΟ και οι συμμετέχουσες χώρες θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στην εκπαιδευτική αυτή αποστολή το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την αφοσίωσή μας στην προσπάθεια που γίνεται στο Αφγανιστάν. Υπενθύμησα στο Συμβούλιο ότι εγώ επισκέφθηκα την Κεντρική Ασία για να συζητήσω με τις χώρες αυτές, όχι μόνο τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, αλλά και ειδικότερα το θέμα του Αφγανιστάν έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο στον τομέα της ασφάλειας της αμοιβαίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και έχουν σαν κομβικό στόχο αν θέλετε την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Προσκαλέσαμε και τον Πίμπαλξ εκεί γιατί πιστεύουμε ότι έχει σημασία να δούμε και συνολικά σφαιρικά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και στον τομέα της ανάπτυξης και συνεργασίας και νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια στρατηγική για τη χώρα αυτή για μετά το 2014. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που τα πράγματα προχωρούν βέβαια, αλλά δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια στιγμή που εμείς έχουμε αποσυνδεθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε να επιδείξουμε κάποιες επιτυχίες, αλλά όπως είδατε όλοι, μέσα στα τα γεγονότα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να πράξουμε, μεταξύ των οποίων και η προετοιμασία των εκλογών για του χρόνου. Είχαμε και μια ευρύτερη συζήτηση στη συνέχεια για την νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολούθησε η διανομή του εγγράφου της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που παρουσιάζει τα μέχρι στιγμή πεπραγμένα και αναφέρει το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να αναφέρω στα μέλη του Κοινοβουλίου πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας στην γειτονιά της Ευρώπης και πιστεύω πράγματι ότι θα πρέπει να έχουμε μια μακροχρόνια δέσμευση, όχι μόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή αυτή. Νομίζω ότι αυτό υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση και τονίστηκε το πόσο σημαντικό είναι όταν εμείς επιδιώκουμε πρόοδο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με υποστηρικτικό τρόπο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει και η συνειδητοποίηση ότι το έργο μας έχει αναγνωριστεί από πολλές από αυτές τις χώρες, από την κοινωνία των πολιτών. Οι προσπάθειές μας να μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τις, ε, σε εμβριακή μορφές, μορφή δομές της κοινωνίας των πολιτών, να δώσουμε φωνή στις γυναίκες, να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε περισσότερο στο να εξασφαλίσουμε να στηρίξουμε τις τόσο εύθραυστες δημοκρατίες των χωρών αυτών να γίνουν πιο αποτελεσματικέ. Φυσικά η Συρία παραμένει, παραμένει πάντα στην καρδιά των σκέψεών μας και έχουμε υπογραμμίσει και πάλι τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για να συγκαλέσουμε τη συνδιάσκεψη Γενέβη 2 για τα θέματα αυτά. Ο εκπρόσωπός μου έχει συναντηθεί με τον κύριο Μπραχίμη, τότε που ήμουν στην Αίγυπτο μίλησα με, τους, με μέλη της ομάδας του. Προσπαθούμε κάθε μέρα να υποστηρίξουμε τη σύγκληση αυτή τη ε, συνδιάσκεψης τη Γενέβη 2 ω απαρχή μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεταβατική κυβέρνηση με πλήρε εκτελεστικέ εξουσίε στη Συρία. <clears throat> Επιπλέον όμω, παραμένει ένα σημαντικό θέμα ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει ανάγκη για μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ιορδανία επισκέφτηκα ε, καταβλισμούς προσφύγων και επίσης και στο Λίβανο. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να μπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να δώσουμε υποστήριξη και είδατε ότι ως αντιπρόεδρος της ε, Κομισιόν μαζί με τον Πρόεδρο κάναμε μια συνάντηση για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν 400 εκατομμύρια περαιτέρω σε απάντηση στην τελευταία έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ. Δεν θα φτάσουν όμως αυτά τα 400 εκατομμύρια. Οι συνέπειες αυτού του τρομερού πολέμου θα πρέπει να μας οδηγήσουν να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση <clears throat> της Συρίας που από όλες τις εκθέσεις φαίνεται ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να υπάρξει υποστήριξη της ανοικοδόμησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς επίσης αναθεωρήσαμε και την πρόοδο στο διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνα. Θέλω να αποτίσω φοροτιμή στους πρωθυπουργούς και των δύο χωρών για τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο έχουν προχωρήσει σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μιλήσει μαζί τους, έχω κάνει πάνω από 100 ώρες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και επίσης 50 άτομα, 25 από κάθε πλευρά, έχουν ευρεθεί με τις υπηρεσίες μου δουλεύοντας σε ομάδες εργασίας συνεχώς, αδιαλείπτως, παραλήλως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το διάλογο αυτό από μια πρόθεση απλώς να εφαρμοστεί, μια ε, χωρίς επιστροφή διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Μπορούν πια τα άτομα να περνάνε τα τελωνιακά τα όρια, τα τελωνία, τα συνοριακές γραμμές χωρίς προβλήματα. Είναι η πρώτη φορά που μπόρεσε να πάει ο εκπρόσωπος της ε, Πριστίνας στο Βελιγράδι και να μιλήσει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν τώρα γραμμία, γραφεία, <clears throat> τα οποία ε, βρίσκονται στις δικές μας, ε, εστιάζονται στις αντιπροσωπείες μας και τους βοηθούν να εργαστούν αλλά δεν υπήρξε μονάχα η συνάντηση που ανέφερα των Πρωθυπουργών, αλλά υπάρχει και καθημερινή συνάντηση και επαφή σε καθημερινό επίπεδο. Συναντηθήκαν επίση όχι μονάχα μαζί μου, αλλά και στι ΗΠΑ και κάνανε μια κοινή επίσκεψη πρόσφατα στην Αυστρία, κάτι για το οποίο θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Αυστριακή κυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία πιστεύω πια είναι ανεπίστρεπτη, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί και ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, θα πάρει μια στεναρή απόφαση επί τη βάση των προτάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλη την υποστήριξη που έχω πάρει και για τους επένους που έχω πάρει από τη δική σας πλευρά και θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά είναι πραγματικά η προσπάθεια των αρχών της Πριστίνα και του Βελιγραδίου που κάναν μια τεράστια προσπάθεια. Εμείς βοηθήσαμε αλλά αυτοί το επέτυχαν. Παραμένουν πάρα πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμα. Στις 8 Ιουλίου θα συναντηθούμε μαζί τους για να συνεχιστεί το έργο αυτό. Εγώ θα σταματήσω τις προσπάθειές μου μέχρι να έχει περατωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να πράξουμε για να εξασφαλίσουμε ότι σε επίπεδο επιτόπιο υπάρχει κατανόηση αυτή τη διαδικασία. Ό,τι μπορεί να κάνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα καλόδεκτο και από τι δύο πλευρέ. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν θέμα, μια σημαντική εξέλιξη όχι μόνο για αυτού αλλά και για όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεχίζω λοιπόν να ζητώ από του Υπουργού Εξωτερικών να υποστηρίξουν τις διμερείς επαφές μεταξύ Κωσόβου και Σερβίας και χαίρομαι που το έχουν πράξει. Ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο θα είναι σαφές τις αποφάσεις τις οποίες θα καταλήξει. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι σας έχω δώσει μια καλή επισκόπηση των ε, συζητήσεων του Συμβουλίου και των αποφάσεων του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την αναφορά σας. Έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές. Θα πρότεινα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων να έχουν 2,5 λεπτά και οι λοιποί 1,5. Αν συμφωνήσετε, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να πάρουν το λόγο. Και είπατε εκπρόσωπος θα έχει την ουσιαστική ευκαιρία να δώσει καλές ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο. Πριν αναφερθώ στα πεπραγμένα του Συμβουλίου, θέλω να εκφράσω μια ανησυχία. Ανα, αναφέρεται αυτή η ανησυχία στα στοιχεία τα αριθμητικά που παρουσίασε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι για την πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2014 σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, όπου παρουσιάζεται μια σημαντική μείωση των κονδυλίων του ύψους των 12,5%. Είναι το πρώτο έτος των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ ελπίζω ο συζητητής της Επιτροπής μας για τα θέματα του προϋπολογισμού να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε με τους κοιόδη συζητητέ αυτή τη δυσκολία. Έχουμε εκφράσει τον πρόεδρο της Επιτροπής προϋπολογισμών την ανησυχία μας για την πρόταση της Κομισιόν. Ελπίζουμε ότι στο, στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση για τα θέματα αυτά των δημοσιονομικών προοπτικών. Έρχομαι τώρα στα τα θέματα που αναφέρατε για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Τρεις ερωτήσεις. Μιλήσατε για την επίσκεψή σας στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο κύριος ε, Κέρι είναι στη Μέση Ανατολή, είναι η πέμπτη του επίσκεψη σήμερα στην Ιερουσαλ... στο Τελαβίβ και την Ιερουσαλήμ, αύριο στην Ιορδανία. Δεν υπήρξαν τώρα σημαντικά συμπεράσματα στο Συμβούλιο Πρόγων Εξωτερικών πέραν της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ερώτημά μας είναι πώς βλέπετε την ε, βιωσιμότητα του σχεδίου που παρουσίασαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τι προσπάθειε αυτέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερο θέμα, η Συρία. Όλοι θέλουμε να γίνει το ταχύτερο δυνατόν η Γενέβη 2, η συνδιάσκεψη αυτή. Δεν φαίνεται ότι αυτό θα καταστεί δυνατό μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχουμε πάνω από 10.000 νεκρούς. Δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα θα υπάρξουν μέχρι τότε. Και δύο ερωτήματα σε σχέση με αυτήν τη συνδιάσκεψη, τη Γενέβη 2. Συζητήσαμε προηγουμένως από εσά με την Χέλγα Σμιτ στο φως των νέων ε, της εκλογής του νέου Προέδρου στο Ιράν. Θεωρείτε ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και τι λέγεται στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, συμπερίληψη των Χεσμολά στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Τέλος, Αίγυπτο, μιλήσατε για τις διαδηλώσεις της 30 του μηνός. Ποιες είναι οι εγγυήσεις που έχετε πάρει για τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης μετά από την ε, προκήρυξη του νέου εκλογικού νόμου για τις εκλογές. Ποιες είναι οι που έχετε πάρει από την κυβέρνηση εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόμις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέιδη Άστον, καλωσορίσατε. Σημερίζομαι τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις σε σχέση με το κομμάτι που αφορά στην υπηρεσία εξωτερική δράση του στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρώτη μου ερώτηση σχετίζεται με το Ισραήλ. Ε, το, Υπουργείο, το Συμβούλιο Εξωτερικών δεν κατέφερε τελικά να εγκρίνει συμπεράσματα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και βάση αναφορών στα ΜΜΕ, στο Ισραήλ και αλλού. θα έχετε επικριτική θέση σε σχέση με τους Ισραηλινούς επικισμούς και την κατεδάφιση ε, Παλαιστινιακών ε, σπιτιών. Μετά από το εντατικό λόμπι, κυρίως ε, του κυρίου Νετανιάχου, διαψέστε το παρακαλώ και εξηγήστε μας για ποιο λόγο ισχύει. Αν ισχύει, ελπίζω πάντως να μην ισχύει. Εμείς γιατί σιωπούμε δε για αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Εσχάτως είδαμε μία δήλωσή σας σε σχέση με την πρόταση του Υπουργού Κέρι και έλεγε ότι δεν ξέρουμε και ότι όταν ξέρουμε τελικά θα τον υποστηρίξουμε. Μα η δική μας η θέση ποια είναι, ανέκαθεν είχαμε θέση, ποια είναι αυτή και πρέπει να την τονίζουμε επανειλημμένα παρότι όντω θα θέλαμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς γιατί θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί να συνασπιστούμε. Γιατί η Συρία Εχθές ε, ε κάναμε μία σύσκεψη, είδαμε διάφορους πολιτικούς χρωματισμούς ε, και είναι πόλεμος ε, δι' αντιπροσώπου και ένα από τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη είναι το Ιράν και είπα στην κυρία Σμιτ ότι το Ιράν θα έπρεπε μέσα στη διάσκεψη της Γενέβης ή ως οποιοδήποτε άλλο φόρουμ να εμπλακεί, διότι έχει σημασία όχι μόνο για τη Συρία αλλά και για το Αφγανιστάν και ξέρετε ποιες είναι οι ανησυχίες μας για το Αφγανιστάν και η Ρωσία επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μας εκβιάζει, μας προκαλεί. Θα ήθελα τελικά να μιλήσω για τη Δυτική Σαχάρα. Την περασμένη, το περασμένο Σαββατοκύριακο ε, κάναμε μια αποστολή στη Ραμπά και στο Ελαγιούν. Δεν θα ήταν αυτό δυνατό αν ε, δεν προχωρούσε τώρα η δημοκρατική τη διαδικασία στο Μαρόκο. Δημοσιεύσαμε μία δήλωση σε σχέση με με τα μέτρα ασφαλείας, ζητούν αυτοδιάθεση οι άνθρωποι και σε σχέση με αυτό που θα γίνουν στην Αλγερία με την εξαφάνιση του Πρόεδρου Μπουτέφλικα, ε, υπάρχει μία πρόθεση των πολιτικών κομμάτων να εμπλακούν σε μία ειρηνική διαπραγματευτική διαδικασία. Τα κάποια κράτη-μέλη μπλόκαραν μία δήλωση ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας σε σχέση με τις εμειονότητες. Ε, διέκοψε ο πρόεδρος την κυρία Γκόμες. Ε, είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σας κυρία Γκόμες λέει. Κύριος Κατσίν, ευχαριστώ. Λίδια στον εξ ονόματος όλων των πολιτικών ομάδων σας καλώ και πάλι να προωθήσετε μια εξισορροπημένη στάση σε σχέση με το θέμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε με, να τηρούμε παθητική στάση όταν ε, ε χιλιάδες ε, χάνουν τη ζωή τους ε, και ξαναρχίζει αυτός ο φαύλος κύκλος των συγκρούσεων ανάμεσα στις θρησκευτικέ κοινότητες. Δεν μπορούμε να έχουμε νέα Βοσνία και εμείς να παρακολουθούμε. Οι χειρότερες ομότητες γίνονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών καλοκαιρινών διακοπών, διότι όλοι αποτιμούν ότι κανεί δεν θα είναι στο γραφείο του για να αντιδράσει, να εμποδίσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θυμηθείτε τη Στρεμπρένιτσα, ε, η σφαγή τότε έγινε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ε, διακοπών. Πεθαίνουν τα παιδιά στου καταβλισμούς προσφύγων, δεν έχουν τα φάρμακα, πεθαίνουν χιλιάδες κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν με τριοπαθείς δυνάμεις που αντιπαλεύουν το δικτάτορο που δεν δείχνει καμία πρόθεση να φύγει από αυτή την αιματηρή οδό που ακολουθεί, Πώς εσείς θα αντιδράσετε σε σχέση με αυτό το κατεπήγον ζήτημα. Δεύτερο θέμα, η Τουρκία. Πρέπει να καταδικάσουμε την απολυταρχική αντίδραση του Ερδογάν ενώπιν μια ειρηνευτική διαδικασία. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να εντάξουμε αυτό το θέμα στη διαδικασία σύνδεση. Είναι ζωτικό συμφέρον για μα. Οι Τούρκοι πολίτε πρέπει να ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ τη ανοιχτή κοινωνία και τη δημοκρατία, όχι μόνο επί τη αρχή, αλλά και στον πραγματικό κόσμο, ακόμη και αν αυτό θέσει εν κινδύνο τι σχέσει μα με στρατηγικό εταιρό, όπω παραδείγματο χάρη η Τουρκία. Ε, ποια είναι η στάση σας και η πολιτική σας και του Επιτρόπου Φίλε για τις ε, τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις. Ε, κατόπιν είμαι εισηγητής για τη Σερβία και θέλω να σας συγχαρώ. Ήταν δύσκολο το έργο σας και στο διάλογο Βελιγραδίου-Πριστίνα έχετε εργαστεί με εξαιρετικό τρόπο. Ο Πρωθυπουργό Κωσυφοπεδίου έδειξε δε ότι έχει ένα πολιτικό όραμα. Θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις του Επιτρόπου Φίλου και της δικής σας για να αρχίσουμε τις, τη διαδικασία σύνδεση με τη Σερβία. Ε, σε σχέση όμως με την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Ε, ξέρω ότι προσπαθεί ο πιο επιρέλη να κάνει ό,τι είναι περνάει από το χέρι του, αλλά αυτή τη στιγμή ε, μία, θα διευκόλυνε, αν σημειωνόταν πρόοδο σε αυτό το ζήτημα, θα διευκόλυνε τη λήψη απόφαση σήμερα ή αύριο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Άστον και τον κύριο Βημό. Δύο ζητήματα, Συρία και Αίγυπτος. Για τη Συρία είναι καλά νέα που τώρα επιτέλους έχουμε μια αντίληψη για το θέμα. Δύο ζητήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να γίνει η διάσκεψη της Γενέβης τι θα κάνουμε με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Ε, μάθατε ότι στο Κατάρ είναι, ε, ο διάδοχος ανέλαβε. Ε, υποτίθεται ότι είναι στο δικό μας στρατόπεδο το Κατάρ. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει υπέρ μας αυτό στις διαπραγματεύσεις για τη Συρία στις απελευθερωμένες περιοχές. Τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω είναι σημαντικό να κάνουμε περισσότερα στο βορρά και στις κουρδικές ε, ε, περιοχές, ελεγχόμενες από τους Κούρδους δηλαδή, γιατί ε, πρέπει να συνεχίσει η καθημερινή ζωή πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι δωρητές του κόλπου όμως δεν μας βοηθούν σε αυτό. Έχουμε έναν μόνο επιτόπο αντί για 15. φυσικά δεν υπάρχει η στελέχωση. Αίγυπτος τώρα. Όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ, ανησυχώ για την, ε, το συλλαλητήριο. Εδώ και εβδομάδες οργανώνεται η διαδήλωση για τις 30 ε, του μήνα και έχουν χαίρε, ε, γιατί παρεμβήκατε κι εσείς, επιμένει να διώκει τους βασικούς εκπροσώπους του τύπου. Δεν είναι πολύ ευφυές εκ μέρους του και επίσης δείχνει ότι είναι εντελώ αυθαίρετη η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα και νιώθουν όλοι ανίσχυροι ως εκ τούτου και άρα κατεβαίνουν όλοι στον δρόμο και ζητούν ε, επανάσταση. Εγώ φόλη φοβάμαι ότι θα επικρατήσει βία και ε, θα πρέπει ρητά να ζητήσουμε ε, ειρηνευτική διαδήλωση αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιος τους χρηματοδοτεί, γιατί καλές οι δηλώσεις, ε, αλλά που πρέπει εμείς να παρακολουθούμε, να καλύπτουμε το συλλαλητήριο, ούτως ώστε να μην αποδοθούν ευθύνες στους νέους για τη βία που μπορεί να μην πηγάζει από αυτούς ή ακόμη και αν πηγάζει από αυτούς δεν θα πρέπει όμως να τους καταγγέλει και να τιμωρούνται ε, Πρέπει να σταματήσει η επιλεκτική δικαιοσύνη, η καταστολή των προσωπικών ελευθεριών. Είναι απαράδεκτο αυτό και να δώσει κάποια σημάδια ε, βούληση σε ε, συνεργασία με την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, παρότι το ζητάμε εδώ και καιρό, δεν υπάρχει. Είναι ε, επίγουσα δε η ανάγκη να συγκροτηθεί μια τέτοια. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπο, πως θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τομή που επιτύγατε στο διάλογο Χριστίνας Βελιγραδίου. Σχετικά με το Μεσανατολικό πράγματι δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει λαμπρές αναμνήσεις σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από διάφορες πλευρές όπως και η ατυχή σας αραβική πρωτοβουλία. Τώρα για τη Μολδαβία υπάρχουν κάποια θετικά βήματα. Για την Ουκρανία υπάρχει φόβος για το αν θα συλλεγούν οι υπογραφές οι οποίες ε, θεωρούν, ε, απαιτούνται. Αναφερθήκατε επίσης ε, και για τη συνάντηση κορυφής στο Μπρουνέι για την ΑΣΕΑΝ. Τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα ανάμεσα στην Κίνα και στην Ιαπωνία για μια σειρά συστάδων νήσων. Ε, τι, πώς θα απορροφηθεί αυτό από το ΑΣΕΑΝ. Επίσης ε, καλό θα ήταν να μπορέσει και η Ταϊβάν να προχωρήσει σε μια σύναψη εμπορικής συμφωνίας με, τις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην συνεχίσει να εξαρτάται απόλυτα οικονομικά από την Κίνα. Τώρα για την Αίγυπτο ε, δημοσιεύθηκε από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου μια καταδικαστική ουσιαστικά έκθεση για την βοήθεια που δίδουμε στη χώρα αυτό. Ε, για την Συρία από ό,τι φαίνεται ο Ασάντ έχει αρχίσει και κερδίζει οπότε γιατί ε, να κάνουμε παραχωρήσεις προς την πλευρά αυτή και καλό θα είναι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο τον Ασάντ έτσι ώστε να αποχωρήσει. Τώρα, σχετικά με τη συμπερίληψη του Χεσμολά στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Από ό,τι μαθαίνω, σε μία από τις χώρες με στη Γερμανία, το Χεσμολά κάνει έρανο για τα έξοδα πολέμου του. Πράγματι, θέσατε πάρα πολλά θέματα ταυτόχρονα και θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε όλα αυτά. Για τον κύριο Σαλαφράνκα για αυτό το ποσοστό το 2,5. Πράγματι ένα τμήμα έχει αλλάξει για τον τρόπο που βλέπουμε εμείς ε, τη στήριξή μας προς ορισμένες χώρες. Κάποιες χώρες έχουν γίνει πιο πλούσιες, έχουν ενισχυθεί οικονομικά και δεν χρειάζονται την αναπτυξιακή βοήθεια όπως ε, την δίδαμε στο παρελθόν. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί υποσυζήτηση και θα συνεχιστεί να συζητάτε στο μέλλον. Ε, δεν ήμουνα στην τέταρτη επίσκεψή μου στην Μέση Ανατολή. Είναι η δέκατη τρίτη επίσκεψη που κάνω στην περιοχή. Η τέταρτη ήταν στη Λωρίδα της Γάζα. Τώρα για το αν το νέο σχέδιο θα είναι βιώσιμο δεν ξέρω. Γνωρίζουμε τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από το σχέδιο αυτό. Το θέμα το οποίο τίθεται ξεκάθαρα είναι το τι μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί για να ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να νιώσουν άνετα έτσι ώστε να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις. Όπως είπα εμείς και σε πολιτικό επίπεδο έχοντας ξεκάθαρες θέσεις αλλά και οικονομικά επειδή είμαστε η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια χώρα του Παλαιστινιακού λαού οικονομικά έχουμε κάνει αρκετά και μπορούμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερο όχι απλά να περιοριστούμε στη συνέχιση της στήριξης αυτής αλλά σε ένα πιο άμεσο θα έλεγα εμπορικό τρόπο και τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ε, να εμπλακούμε ακόμα περισσότερο μαζί τους. Τώρα, <clears throat> στις συναντήσεις στη Γενέβη προφανώς θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ιρανοί. Έχουν τεθεί πολλά θέματα εδώ και το θέμα της Συρίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει κανείς. Θα πρέπει να δούμε τι κυβέρνηση θα έχουμε στο Ιράν. Για κάποιους πιστεύουν ότι ε, αν ξεχωρίσουμε το θέμα του Ιράν από τη Συρία δεν θα έχουμε προοδεύσει σε κανένα από τα δύο θέματα. Γιατί με τον ένα τρόπο ή τον άλλο εμπλέκονται. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε και μέσω των Ηνωμένων Εθνών ε, να πιέσουμε τους Ιρανούς έτσι ώστε να δούμε με ποιους θέλουν εν πάση περιπτώσει να διαπραγματευθούν. Και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτών όλοι όσοι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, στην περιφέρεια αυτή, στην περιοχή καλύτερα αυτή, να μην είναι απόντες. Εδώ ακούγονται πολλές χώρες, ακούγονται πολλές ομαδοποιήσεις χωρών. Θα πρέπει όλοι αυτοί να καταλάβουν ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και ότι η διαδικασία αυτή οδεύει προς μια κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να αποδεχθούν για να συνεισφέρουν στο να ξεπεραστεί το θέμα, αντιμετωπιστεί το θέμα. Για το Χεσμολά. Έχω θέσει το θέμα επανειλημμένα και στο θέμα εξωτερικών υποθέσεων και στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Η απόφαση αν ληφθεί όταν ληφθεί πρέπει να είναι ομόφωνη και υπάρχουν δισταγμοί και διαφορές. Όχι ότι δεν ανησυχούν οι χώρες μέλη, αλλά σχετικά με το θέμα του Λιβάνου σαν παράδειγμα πόσο αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Λίβανο το να συμπεριλάβουμε την οργάνωση αυτή σε τρομοκρατική λίστα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά να εξετάζουμε. Εγώ επισκέφθηκα και τα στρατεύματα που έχουμε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ <clears throat> και με ενημέρωσε ο στρατιωτικός διοικητής των στρατευμάτων αυτών που κάνουν τεράστιες προσπάθειες σε μια κατάσταση η οποία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Τώρα, για την Αίγυπτο ε, θα επανέλθουμε αργότερα στα θέματα των διαδηλώσεων κτλ. Αλλά εγώ όταν έφυγα από την Αίγυπτο την τελευταία εβδομάδα ήμουνα πολύ ανήσυχος. Εγώ συναντήθηκα με αντιπολιτευτικά κόμματα, με ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών Είχα πολύ ενδιαφέρουσες και μακρότατες συζητήσεις, αλλά ανησυχώ για το τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι <clears throat> πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε οι διαδηλώσεις να διεξάγονται ειρηνικά. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν οι διαδηλώσεις αυτές να διεξάγονται με ειρηνικό τρόπο Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, χωρίς φυσικά να εκθέτουμε σε κίνδυνο τους ανθρώπους μας στη χώρα αυτή. Ακούγονται φωνές και όταν ήμουν εκεί που θέλουν να βρεθούν πραγματικές λύσεις. Η δημοκρατία δεν είναι το να εκλεγεί κάποιος κάπου, το θέμα είναι τι κάνει αυτή τη στιγμή σε εκλεγεί. Η δημοκρατία είναι μια ολόκληρη σειρά από αριθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε ο λαός να νιώσει ότι η ζωή του αλλάζει, ότι συμμετέχει, ότι ακούγεται, ότι η κοινωνία των πολιτών παίζει ρόλο στο σύνολο της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ανήσυχη για την Αίγυπτο, ε, γενικά ανησυχώ για την Αίγυπτο, πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό Αυτά θα τα συζητήσουμε πάλι και σε διμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις γειτονικές της Αιγύπτου χώρες. Για τα συμπεράσματα δεν ε, νομίζω ότι αποτύχαμε εμεί τις προσπάθειες που κάναμε εκεί. Το τι λένε τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ έχει πάψει να με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό ακριβώς το είπα στο Συμβούλιο. Έχει μεγάλη σημασία να ανοίξουμε κάποιες προοπτικές και με ενεθάρρυνε αυτό το οποίο άκουσα στη Ραμάλα και στη Δυτική Όχθη. Μπορεί να υπάρξει πρόοδος και πρέπει να στηρίξουμε την πρόοδο αυτή τη νέα διαδικασία. Δεν είμαστε μόνο λόγια. Εμείς πιστεύουμε αυτά τα οποία λέμε. δεν έχω αλλάξει την άποψή μου για τις ε, εγκαταστάσεις ας πούμε των επίκων. Είναι παράνομες και εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι παράνομες. Ανησυχώ λοιπόν για κάποια πράγματα που γίνονται στη περιοχή αυτή και το ξεκαθάρισα στους Ισραηλινούς, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στους εκπροσώπους του στη Δυτική Όχθη. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνουν βήματα προόδου πάντως στην παρούσα φάση και είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Κέρι αποφάσισε να αφιερώσει την ενέργειά του στον τομέα αυτό, στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχει εμπειρία, έχει στήριξη, έχει επιμελητία και μεγάλη υψηλή αξιοπιστία και μπορεί να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον κόσμο να εμπλακεί σε κάποια μορφή διαπραγματεύσεων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μου το ξεκαθάρισε ο Υπουργό Κέρι είναι πολύτιμη στη διαδικασία αυτή και γι' αυτό του είπα ότι θα τον στηρίξουμε και το Συμβούλιο επίσης. Θα πρέπει φυσικά να γίνουν περισσότερες συζητήσεις, αλλά αποφασίσαμε ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε στην παρούσα φάση ότι στηρίζουμε τις προσπάθειές του. Έκανα όμως σαφές ότι, και το είπα αυτό και στον, στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον τότε πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και τον πρόεδρο Μαχμού Ταμπάς, ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες μας. Τα μέσα ενημέρωση γράφουν πάντα αυτό που θέλουν. Αυτό δεν εκπλήσει κανένα. Για τη Συρία τώρα θέσατε το ερώτημα για, την, για το ρόλο του Ιράν. Και αυτό που είπατε για το Αφγανιστάν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Ένα από τα πράγματα που λέμε στου Ιρανούς είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του Αφγανιστάν. Είναι ένα κοινό θέμα για όλου μα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα για την ε, συμμετοχή του Ιράν στα θέματα αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι να εξασφαλίσουμε ότι αν υπάρχει μια καλή διαδικασία, ότι όλοι θα νιώθουν δεσμευμένοι να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια για να υπάρξει ένα ομαλό μέλλον στη Συρία και ένα μέλλον για το λαό του, του Συριακού λαού, δηλαδή να μπορέσουν να δεσμευτούν όλες τις προσπάθειές τους για τη Δυτική Σαχάρα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είναι και συμβιβαστική τελικά κατάσταση για λόγους που ξέρετε πολύ καλά Προσπαθούμε να καταφέρουμε να προχωρήσουν οι προσπάθειες του ΟΗΕ και του Μπανκιμούν στο βαθμό του δυνατού. Και το ίδιο πράγμα <clears throat> κάνουμε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική λύση. Απλώς λοιπόν εδώ υποστηρίζουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον ΟΗΕ. Κάποιες φορές προσπαθούμε να τους ε, σπρώξουμε, άλλες φορές στεκόμαστε δίπλα τους και τους υποστηρίζουμε απόλυτα στις προσπαθίες τους. Κύριε Κάτσιν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που αναφέρατε για αυτά που κάνουμε στην Σερβία, θα επανέλθω σε αυτό, για την ε, Συρία, για το να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για τη Συρία. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο συζήτησε επί 12 ώρες για να μπορέσει να καταλήξει σε μια θέση η οποία θα επιτυγχάνει αυτή την ισορροπημένη θέση. Καταρχήν όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να βρεθεί μια πολιτική διαδικασία για να επιληθεί τώρα η κατάσταση στη Συρία. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε αυτή την πολιτική διαδικασία, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσουν οι μάχες. Αλλά υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και έγκυρες απόψεις για το πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να μπορέσουμε να δείξουμε με ορατό τρόπο υποστήριξη προς τους ε, αντιμαχόμενους των Άσαντ. Λένε ότι πρέπει να δώσουμε όπλα, άλλοι λένε στους, ε, σε αυτούς. Άλλοι λένε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κλιμάκωση γιατί θα οδηγήσει σε περισσότερα όπλα και προς τον Ασάντ και θα αυξηθούν οι συγκρούσεις. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να καταλήξουν σε μια πολιτική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει εν καιρό σε μια λύση που θα φέρει μόνιμη ειρήνη στη Συρία. Όλες μου οι προσπάθειες λοιπόν κατευθύνονται προς τα εκεί. Τα κράτη-μέλη πήραν μια απόφαση μετά από μακρές συζητήσεις, θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα να μπορεί να δίνει κανείς όπλα στην αντιπολίτευση του Ασάντ μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν στοιχείο των συζητήσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Τώρα είναι στο χέρι των κρατών μελών να προχωρήσουν ή να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και η ομάδα σα είναι σίγουρα μέσα σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια πολιτική διαδικασία. Δεν θεωρώ και εγώ ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό πολύ γρήγορα. Πρέπει να γίνει όμως σύντομα, το ταχύτερο που θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό τόσο το καλύτερο. Ε, στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάει στην ανθρωπιστική βοήθεια και εξακολουθούμε να, δου, να <clears throat> κοιτάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και εδώ πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια πολιτική διαδικασία στη Συρία. Για την Τουρκία. Ρωτάτε τι κάνουμε. Υπάρχει πάντα αυτό το φάσμα μεταξύ μιας ε, ενεργητικής στάσης και της απομόνωσης της Τουρκίας. Εμείς μένουμε σε επίπεδο επαφής με την Τουρκία και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την επαφή, να στέλνουμε ισχυρά μηνύματα, να συνεχίσουμε να είμαστε σαφείς για τη θέση μας, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ σαφέ ότι ο λαό της ε, Τουρκίας θέλει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία και θέλει την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κομμάτι της ε, Πορεία τη Τουρκία στο μέλλον. Αυτή είναι και η δική μου προσωπική άποψη ότι πρέπει η Τουρκία να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για αυτού και για μας. Για την Σερβία, για την ενέργεια και την ε, ε τηλεπικοινωνίες. Έχει πια ένα αριθμό στο διεθνέ τηλεφωνικό δίκτυο, το Κωσυφοπέδιο που είναι το 315. Οι ομάδε εργασία συνεχίζουν να εργάζονται για τα θέματα αυτά. Τα θέματα τηλεπικοινωνιών έχουν περίπου περατωθεί. Είναι δύσκολο βέβαια όταν κάποιοι δεν αναγνωρίζουν αυτή τη χώρα ως οντότητα. Είναι δύσκολο να μπορεί να έχει ένα τηλεφωνικό αριθμό και έχουμε κάποια προβλήματα. Για το θέμα της ενέργειας υπάρχει σημαντική πρόοδος και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά πράγματι είναι δύσκολα τα θέματα αυτά. Κυρία Μπραντνερ. Είπα κάποια πράγματα ήδη για τη Συρία και για τη σημασία που έχει το να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στην αντιπολίτευση. Συνεργαζόμαστε στενά και υπάρχει μονίμως κάποιος το Γατζιαντέπ Έχουμε ανθρώπους από την ΕΚΟ και από την ΤΕΦΚΟ, της Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή. Ε, κάνουμε προσπάθειες. Ε, μας μιλήσατε για το Κατάρ και τις αλλαγές. Ε, την, ε, έχουμε τη σύσκεψη με τα κράτη του κόλπου το Σαββατοκύριακο και εγώ θα παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τις αλλαγές και θα προβληματιστούμε για το τι συμβαίνει εκεί. έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει το ζήτημα και το Σάββατο και την Κυριακή θα πάω στο Μπαχρέιν, πρωτού πάω στο Πρινέ γιατί προεδρεύω στη σύσκεψη. Για την Αίγυπτο ε, μιλήσαμε πάρα πολύ εκτεταμένα με τον Πρόεδρο, τα είπα όλα αυτά, η, κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δέσμευση και αφοσίωση που πρέπει να δείξει, η ανάπτυξη δεσμών με την αντιπολίτευση, το συμφέρον της χώρας είναι ε, το υπέρτατο ζητούμενο και τα όσα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες έχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Ε, Του μίλησα για τις ανησυχίες σε σχέση με το διορισμό κυβερνητών ε, επίσης για το ότι δεν ισούται η εκλογική διαδικασία με τη δημοκρατία. Είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας και οφείλω να πω ότι συζήτησε ουσιαστικά μαζί μου ε, βεβαίως δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουν οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά εκεί θα είναι, θα παρακολουθούν τη διαδικασία και θα υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών. Θα απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση ε, να ακουστούν όλες οι φωνές ε, με ήπιο τρόπο. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και ελπίζω να διαπιστώσουμε ότι έτσι συνέβη την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με την λαϊκή δυσαρέσκεια. Κύριε Τάνοκ, για την Ουκρανία Ευχαριστώ για, τα, για τις φιλοφρονήσεις σας για τη Σερβία. Ελπίζω, ελπίζω να πετύχω τα ίδια και στη Μέση Ανατολή. Αυτά που είπατε για τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο αποδεικνύουν το τι μπορούμε να κάνουμε ε, και στο μέλλον. Ε, ελπίζω να μην είναι το μόνο και αυτά που κάνουμε στη Σομαλία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή πράγματα ε, που κάνουμε στην γειτονική περιοχή αποδεικνύουν το δυναμικό της κοινή δράσης. Δεν μπορούμε να δρούμε μονομένα. Ε, τώρα δίκιο έχετε, άμα το πάρουμε την υπογραφή, τι μήνυμα θα περάσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιε είναι οι δικέ μα οι προθέσει, αλλά επίση να ξεκαθαρίσουμε ότι θα κάνουν και εκείνοι αυτό που του αναλογεί. Ε, και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το σύστημα επιλεκτικής δικαιοσύνης και δικαστικών μεταρρυθμίσεων ε, και παρενθετικά να πω ότι ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν αλλά στη συνάντηση της Δευτέρας ε, με τον Πρόεδρο γιατί με τον Επίτροπο Φίλε συναντηθήκαμε σύντομα μαζί του και ξεκαθαρίσαμε όλα αυτά τα σημεία και ελπίζω ότι τελικά θα είναι σε θέση η κυβέρνηση να τα τα κάνει αυτά, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ελπίζουν να το κάνουν. Εμείς πάντως ξεκαθαρίσαμε ε, τη θέση μας ε, και όπως ξέρετε μας ενδιαφέρει το ευρύτερο ζήτημα του ΑΣΕΑΝ ε, και τα εμπορικά θέματα. Θα ήθελα δύο-τρεις παρατηρήσεις να κάνω συγκεκριμένα για αυτά. Εγώ θα ήθελα το ελεγκτικό συνέδριο φυσικά να συντάσει ποιοτικέ εκθέσεις και εν θα συμφωνήσω με την έκθεση πάντως στείλαμε εκτεταμένα σχόλια σε σχέση με το προσχέδιο. Δυστυχώς δεν συμπεριλήφθησαν αυτά τα σχόλια τέσσερα από τα 15 κεφάλαια είναι αρνητικά. Όταν, αν διατρέξετε όμως την έκθεση θα δείτε ότι είναι μάλλον θετικό το κλίμα. Ε, μιλάμε για την περίοδο μέχρι το 2012. Αν μπορούμε να λύσουμε διδάγματα. Γι' αυτό έχουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Μας υποδεικνύει τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. θα προτιμούσα και εγώ μια διαφορετική παρουσίαση των ζητημάτων. Υπάρχουν ε, αναρρύθμιτα δημοσιεύματα στον τύπο και μιλάνε για δισεκατομμύρια ευρώ ε, που δαπανάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδρομή 40 εκατομμύρια είναι αυτά. 900, ε, 960 ε, ε, δεν δαπανώνται από εμά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι χρησιμοποιούμε τα κονδύλια για τι γυναίκε για να έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε υγείας. Υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών, Δράσει για την ανεργία των νέων. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι δράσει. Αυτά εκταμιεύσαμε και στην ομάδα ειδική δράση περιμένουμε το δούνο του. Δεν έχουμε εκταμιεύσει σε τίποτα. Οπότε συμφωνούμε, υπάρχει σύμπνοια με το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ υπεραμείνω με του ε, δικαιώματό του πάντω να απευθύνουν επικρίσει ε, και δεν πρόκειται να αλλάξω στάση. Σα ευχαριστούμε, κυρία Σαΐφ. Κυρία σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Το ερώτημά μου αναφέρεται στο... στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την Αίγυπτο. Μα δώσατε ορισμένα στοιχεία αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ. Τα... Οι μεγάλοι τίτλοι στις εφημερίδες το παρουσίασαν ως κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Ότι δεν είναι αποτελεσματική η υποστήριξη η οποία δίνεται. Ξέρω ότι έχετε κάποια στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσατε, τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί, δεν είχαν παρουσιαστεί από τα μέσα της ενημέρωσης, αλλά η έλλειψη διαφάνειας, ο μη σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών παραμένει. Θεωρείτε ότι τα ίδια σχόλια μπορούν να ισχύουν και για άλλες χώρες της περιοχής και ιδίως αυτή η λογική του περισσότερα για περισσότερα. Αυτό ήταν η κύρια κατεύθυνση της πολιτικής μας. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική μας. Ένα δεύτερο θέμα. Αναφερθήκατε στο Συμβούλιο με τις χώρες του Περσικού Κόλπου στις 30 Ιουνίου Μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για την ημέρηση διάταξη και τις προτεραιότητες αυτής της συνάντησης. Σας ευχαριστώ Λέδη Άστον για την παρουσία σας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ένα θα ήθελα να θέσω, το οποίο θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα. Την δημοκρατική μετάβαση στην Τινησία. Γνωρίζετε ότι η συνταγματική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών υπάρχει αυτή τη στιγμή έλεγχος και σε σχέση με την συντακτική συνέλευση. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή θετικά θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς για το σύνολο της περιοχής. Το κείμενο που έχει συνταχθεί είναι χρήσιμη βάση, αλλά υπάρχουν κάποιες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχουν αρκετά αρνητικά σημεία και το έχει υπογραμμίσει η κοινωνία των πολιτών. Να σας δώσω λίγα παραδείγματα. Περιορίζεται το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης του τύπου, των μέσων ενημέρωσης, η αρχή της αναλογικότητας, ο αρχηγός του κράτους πρέπει να είναι μουσουλμάνος, διευκρινίζεται, οι συνταγματικές εγγυήσει για την ανεξαρτησία του ανεξάρτητου δικαστικού συμβουλίου είναι ανεπαρκής. και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις για τη σχέση που μπορεί να έχει ο πρόεδρος του κράτους με τον Πρωθυπουργό γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις η σχέση αυτή ανάμεσα στους δύο εις βάρος της χώρας. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν για να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο προτινόμενο σύνταγμα υποστηρίζοντας τις ε, προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών. Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε λίγες εβδομάδες και πρέπει να βιαστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, λέει ο κύριος Πέτρινγκ. Ο κύριος Πρόκ αναφέρθηκε στην απόφαση δικαστική κατά τον ιδρυμάτων στην ε, Αίγυπτο, πρέπει να τονίσω ότι αυτό πραγματικά είναι παράλογο. Υπάρχει απουσία ενός κράτους δικαίου. Θα ήθελα να σταθείτε στο θέμα αυτό. Λένε, η, λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαδικασία. Αλλά λέει τώρα δικαιοσύνη πρέπει να εκδοθούν διεθνή ε, εντάλματα σύλληψης. Αυτό σημαίνει ότι τα 43 αυτά εμπλεκόμενα άτομα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό αναφέρεται και στα άτομα που εργάζονται στο Ίδρυμα Conrad Adenauer, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και οι Αμερικανοί, οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το Ίδρυμα και υπάρχει ο γερουσιαστής Μακέν και η κυρία Ολμπράιτ, η πρώην υπουργό Εξωτερικών που συνδέονται με το Ίδρυμα Conrad Adenauer. Λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσετε και εσείς τι σημαίνει αυτή η έκδοση διεθνών εντάλματων συλλήψης για τα άτομα αυτά που εργάζονται εκεί. Και ίσως πρέπει να δείτε πώς αντιμετωπίσετε το θέμα των ε, νόμων για τις ΜΚΟ, όχι μόνο στην Αιγυπτό αλλά και στο Εκουαδό σε σχέση με τη δυνατότητα ΜΚΟ να εργάζονται που είναι περιοριστικό, αλλά και στην Ρωσία. Πρέπει να δείτε πώς αντιμετωπίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που πρέπει να δέχονται να παρουσιάζονται ως ε, ξένοι πράκτορες όταν έχουν επαφές με ρωσικές ε, οργανώσεις. Αυτό πραγματικά είναι μια απειλή προς, τις, ε, προς την κοινωνία των πολιτών και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αν θα το εξετάσετε το θέμα αυτό εντελεχώς και πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ε, κυρία τη εκπρόσωπε, θα ήθελα τις κάποιες διευκρινήσει σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που το ελεκτικό συνέδριο θεώρησε ότι χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο αναποτελεσματικό. Ελέγχθη ότι χρησιμοποίησαμε μόνο 14 εκατομμύρια από το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό δεν μπορεί να στέκεται. Δεν ξέρω αν εσεί μίλησατε για τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν τώρα, θα εκταμιευτούν τώρα. Αλλά το ελεκτικό συνέδριο αναφέρεται σε κονδύλια μεταξύ 2007 και 2012. Είναι πολύ σημαντικό και εσεί και ο Επίτροπος Φίλε να εξηγήσετε καλύτερα τι έγινε. Γιατί αυτό οδηγεί σε τυχαίου τίτλου και δεν είναι ακριβώς οι τίτλοι που θέλουμε να γράφονται για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε μια εποχή κρίση πρέπει να είμαστε υπόλοιποι στου πολίτε μα για το πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα και είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, επομένω απαιτούνται σοβαρέ απαντήσει. Είπατε μετά ότι είναι οι δράσει που μετράνε και όχι οι δηλώσει. Διάβασα όμω μια δήλωση που κάνετε στι 19 Ιουνίου αφού συναντήσατε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Θα ήθελα να ξέρω τι έχετε να πείτε για την πολιτική αυτή του More for More, για την ερεσιμότητα, για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Τίποτα από όλα αυτά δεν αναφερόταν στο, στη δήλωσή σας. Αναρωτιέμαι, σε ποιον απευθύνεται η δήλωσή σας ποιος θα πρέπει να επηρεαστεί από αυτή τη δήλωση και γιατί δεν αντανακλώνται αυτές οι βασικές έννοιες και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστεύω ότι υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των κρατών μελών και από εμά εδώ και που θα πρέπει να γίνουν ακουστές και από το λαό της Αιγύπτου αλλά και από την κυβέρνηση της Αιγύπτου. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέβη Άστον, θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία που σχολιάσατε και γύρατε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Μιλήσατε για τις κλιματικές αλλαγές και τη σχετική στρατηγική. Αυτό επηρεάζει φυσικά και τις μετακινήσεις, τις πληθυσμιακές. Και από όσο ξέρω δεν υπάρχει καμία συνεκτική ε, προσέγγιση για το θέμα των κλιματικών προσφύγων. Στο ανακοινωθέν τύπου δεν είδα καμία αναφορά σε αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να το αιτιολογήσετε. Δεύτερον, Πακιστάν και η Εμένη συζητήθηκε στο Συμβούλιο και στις δύο χώρες ε, μιλάμε για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τη χρήση τους ε, που οδήγησε σε πολλούς ε, θανάτους στους αμάχους. Είχαμε τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξοδικαστικές εκτελέσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε ισχυρή θέση καταδικάζοντας το θέμα των εξοδικαστικών δολοφονιών ε, αναμένεται πολιτικός διάλογος ε, για την αντιτρομοκρατική δράση στο Πακιστάν. Θα το θέσετε το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για αυτό το ζήτημα, ε, διότι υπάρχει και το θέμα της παραβίας του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον. Ως συμπρόεδρο της Euronest θα ήθελα να σας συγχαρώ. όχι μόνο για την προτεραιότητα για την ανατολική εταιρική σχέση και την επερχόμενη σύνοδο του Βίλνιους, αλλά για το ότι είναι κρίσιμη η περίοδος. Είναι πολύ θετικό που θα το θέσετε και ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών Στι στις 22 Ιουλίου στα πλαίσια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι σημαντικό διότι αναφερθήκατε σε αυτό το αίσθημα που πρέπει να έχουν όλοι ότι, είναι, ότι έχουν και οι ίδιοι κινήσει και δρομολογήσει τη διαδικασία να μην θεωρήσουν ότι κάποιος επιβάλλει αξίες και ιδέες. Αυτό όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που με ανησυχεί όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, δεν κάνουμε τίποτα για τις ε, παρατεταμένες συγκρούσεις ε, στην Νότια Οσετία, στην Υπερτινιστερία, στον Αγκόνο Καραμπάχ. Γιατί και εκεί είδαμε λίγα ανησυχητικά σημάδια πρόσφατα. Κατά τη γνώμη μου, για να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας, θα πρέπει να τραβήξουμε περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό, διότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκή επικρατή, είναι άμεση γείτονές μας. Πρέπει να επιδιώξουμε αυξημένη επιρροή σε αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Άστον. Χαίρομαι που πάντοτε όταν σας βλέπω εδώ στην ΑΦΕΤ Βελιγράδη, Πρίστινα και Διάλογος. Ε, επενέσατε δύο πρωθυπουργούς και τα επιτελεία τους. Αντικειμενικά όμως σας πρέπει να συγχαρούμε διότι ο ρόλος σας στη διαδικασία είναι καταλυτικός από την αρχή μέχρι σήμερα. Τώρα τι γίνεται. Αν συμβεί κάτι που δεν θα εκτροχιάσει, ελπίζω, την όλη διαδικασία. Θα ήταν καλύτερο όχι μόνο για τους δύο εταίρους, αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα το έπαιρνα προσωπικά. Τι σας ερωτώ. Τι θα γίνει μετά το πέρας της διαδικασίας. Μιλάμε για εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο εταίρους. Θα δημιουργηθεί μια θετική ενέργεια, αλλά μετά μετά τι θα γίνει, προβλέπετε διάλογο ή άλλη πρωτοβουλία για να επέλθει η τελική λύση για το Κωσυφοπαίδιο στην Αλβανία ε, με τις κοινοβουλευτικέ εκλογές στην Κυριακή στα Τύρανα. Είναι ένα τεστ, ένα πολιτικό πείραμα για την οριμότητα της Αλβανίας, για το λαό και κυρίως για την πολιτική ελίτ της Αλβανίας. Συνεχίζεται αυτό το πείραμα. Ε, ήταν φυσιολογικό το τραγικό δυστύχημα στις εκλογές είναι προοδευτικοί μάλλον οι πολιτικοί ηγέτες. Ας τους βοηθήσουμε να φέρουν σε πέρα σε αυτή την ομαλή μετάβαση ε, και έτσι να αναβαθμίσουμε και αυτή την βαλκανική χώρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι προς τη Λέδη Άστον λέει η κυρία Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με την Τουρκία. Υποστηρίζω την ιδέα να βοηθήσουμε την Τουρκία να προχωρήσει και να στραφεί ακόμα περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέματα που αφορούν και τη Βουλγαρία και αναφέρομαι στα δικαιώματα ιδιοκτησίας αυτών που εγκατέλειψαν την Θράκη και υπήρξε μάλιστα και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και το δεύτερο θέμα μας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί κάπως η στρατηγική. Αναφερόμαστε στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι που παρέχει η περιοχή αυτή. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές αλλαγές στην περιοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με, τις, με τους πόρους από την εκμετάλλευση της ενέργειας που μπορεί να περνάει από την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Για την κυρία Σαϊφή. Αναφερθήκατε στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα θέματα της διαφάνειας και για το εάν αυτά στα πλαίσια της διαδικασίας more for more θα εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον τομέα της διαφάνειας στον τρόπο που λειτουργούμε. Οι εκθέσεις τις οποίες επεξεργαζόμεθα τώρα αφορούν μία περίοδο η οποία αφορούσε θα έλεγα την κατάσταση πριν από τις δραματικές αλλαγές τις οποίες βλέπουμε τώρα πρόσφατα. Αναφερόμαστε δηλαδή σε καθεστώτα τα οποία προσπάθησαν να διασφαλίσουν μία κάποια θετική εξέλιξη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τελικά η ανατροπή αυτών των καθεστώτων έδωσε την δυνατότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν αντικείμενο καλύτερου σεβασμού, όχι όμως καμία διασφάλιση ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντα το χάος ε, ελοχεύει και όταν πήγα στην Ισία ήμουνα η πρώτη διεθνής εκπρόσωπος που μπήκα σε γραφεία οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, εκεί υπήρξε και μια προσπάθεια συντονισμού μεταξύ τους. Η προσπάθειά μας λοιπόν βοηθά γενικότερα την προώθηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και αν κάποιος πιστεύει ότι αυτές οι ταραχές θα οδηγήσουν σε μια θαυμαστή δημοκρατική κατάσταση μέσα σε λίγο καιρό, το Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς την ιστορία θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα και οι απαντήσεις δεν είναι δεδομένες. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα την λύση. Για τη συνάντηση αυτή GCC το Σαββατοκύριακο συζητήσαμε κυρίως δύο θέματα. Πρώτον στις διμερείς σχέσεις μεταξύ μας που καλύπτει και την οικονομία, την ανάπτυξη και τα, τις πιθανότητες ε, υπογραφής μιας εμπορικής συμφωνίας, το θέμα των θεωρήσεων, το οποίο ενδιαφέρει και εσάς σαν κοινοβούλιο, και γενικότερα ευρύτερα περιφερειακά θέματα σε τομείς που, στους οποίους αναφερθήκαμε σήμερα το πρωί. Πάντα στα, όταν συζητάμε με την Αίγυπτο τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπρόσωπός μου είναι στον Μπαχρέιν σήμερα και προετοιμάζει τις συναντήσεις τις οποίες θα έχω από το Σάββατο. Για τον κύριο Παντσέρη, για την Τινησία. Εμείς με ιδιαίτερα τακτό τρόπο πιέζουμε την κυβέρνηση για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει στις συνταγματικές αυτές προτάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Θέσαμε πάρα πολύ δύσκολα θέματα και όταν ήταν εδώ την προηγούμενη Τρίτη ο Πρωθυπουργό, εγώ δεν τον συνάντησα γιατί ήμουν δυστυχώ στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, αλλά συναντήθηκε με τους Προέδρους Μπαρόσο και Βαν Ρομπέι και του πέρασαν ξεκάθαρα μηνύματα και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον κύριο Πέτερινγκ. Πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας για τις ΜΚΟ. Εγώ ξεκίνησα ένα διάλογο με κάποιες κομβικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν περιορίζεται σε μία χώρα ή σε μία περιοχή. Στα πλαίσια της εφαρμογής της αρχής More for More είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις σε σχέση με τις ΜΚΟ σε ορισμένες περιπτώσεις ενώ σε άλλες χώρες ε, ε, έχουν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική. Προσπαθώ λοιπόν να συνδυάσω έτσι ώστε τις προσπάθειες που γίνονται για να βοηθήσουμε συντονισμένα τις ΜΚΟ για τις ορισμένες χώρες όσο πιο ισχυροί είμαστε και ενωμένοι τόσο το καλύτερο γιατί υπάρχουν και χώρες όπου κοιτάνε με πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα το τι μπορεί να κάνουν οι ΜΚΟ και δεν κατανοεί ο κόσμος τις δυνατότητες βοήθειας και ανάπτυξης που έχουν. Δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται τα ωφέλη τα οποία μπορεί να φέρουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα πρέπει να τις συντονίσουμε, να υπάρξει συνένεση για τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα υπερασπιστούμε τις ΜΚΟ, θα στηρίξουμε τη ΜΚΟ σαν μια συνεκτική ομάδα. Γιατί αλλιώς μία προς μία ε, ε, διασπείρουν τις προσπάθειές τους προς κατευθύνσεις όχι εύκολα συντονιστές. Σάκε. Νόμιζα ότι είχα αναφερθεί σε σχέση με το ένα δισευρο. Η έκθεση όπως είπατε αναφέρεται σε ποσά τα οποία είχαν δαπανηθεί στο παρελθόν. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα. Το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει προσεκτικά το τι έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ένα τμήμα αυτής της περίοδου καλύπτει και τη δική μου περίοδο. Πώς έχουν δαπανηθεί οι πόροι τους οποίους είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτή η ελεγκτική διαδικασία είναι εξαιρετική. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να πω είναι ότι τα σχόλια τα οποία εμείς κυκλοφορήσαμε για την έκθεση αυτή δείχνουν πως ποικίλει η κατάσταση από χώρα σε χώρα και κάποια από τα σχόλια αυτά θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου. Παρ' όλα αυτά το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να μην τα δημοσιεύσει. Αυτή είναι η δουλειά του, αυτό αποφάσισε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια σε σημαντικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να χρησιμοποιούμε σωστά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί κανείς τα χρήματά του. Κάποιες χώρες θέλουν στήριξη δημοσιονομική, κάποιες όχι. Κάποιες θέλουν σαν παράδειγμα να χρησιμοποιούνται για υποδομές κυβερνητικές, άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα χρήματά μας εκτός κυβερνητικών δομών στις διάφορες χώρες που παρεμβαίνουμε. Υπάρχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις, η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει με ιστερικό τρόπο και μπροστά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο που λειτουργούμε σε χώρες που σε αυτή την περίπτωση είναι σε αναταραχή ή πριν από κάποια περίοδο αναταραχής ή ακολουθούν αμέσως μια περίοδο αναταραχής. Και αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να εξασφαλίσουμε σταθερότητα, να υποστηρίξουμε το λαό των χωρών αυτών και να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν. Και η λογική περισσότερα για περισσότερα είναι μια πολύ καλή φράση, επινόηση του Στεφάνου Φίλε. Είναι ένας καλός τρόπος να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, αλλά πολλές φορές το, κατά κάποιο τρόπο το, το διαστρεβλώνουν για να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε ότι σε μια ομάδα ε, γυναικών ότι επειδή η κυβέρνησή σας συμπεριφέρετε με άσχημο τρόπο, δεν θα σας δώσουμε καθόλου λεφτά. Όχι. Αντίθετα είπαμε ότι όταν μια κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τις μεταρρυθμίσεις θα τους δώσουμε περισσότερη υποστήριξη. Αυτό σημαίνει το more for more. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε κίνητρα και να βοηθήσουμε να γίνονται περισσότερα πράγματα με το να ξέρουν οι κυβερνήσει ότι αν κινηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Για μένα όμω δεν σημαίνει ότι λέω στι γυναίκε, σε οργανώσει των γυναικών, ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, εμεί θα μειώσουμε τη χρηματοδότησή σα. Ας είμαστε λοιπόν σαφείς, ας σε δώσουμε το σωστό πλαίσιο για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα. Και οι εφημερίδες γράφουν πάντα ό,τι θέλουν. Δεν νομίζω ότι οι ειδήσει στον τύπο για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αντανακλούν την πραγματικότητα. Εγώ είμαι ευγνώμων για το ελεκτικό συνέδριο που μας είπε όλα αυτά τα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έρχεται κάποιος από 500 δηλώσεις μία δήλωση και λέει αυτή τη δήλωση δεν χρησιμοποίησα τις λέξεις που θέλατε να χρησιμοποιήσω. Μπορώ να σας βρω άλλες 50 ε, δηλώσεις όπου τις χρησιμοποίησα. Αλλά δεν μπορώ να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο ότι στην τάδε δήλωση εγώ δεν έκανα τις ε, απαραίτητες ε, δεν είπα τις απαραίτητες φράσεις στην Αίγυπτο στη συνάντηση με τον Χαμαντιάμπα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνω πιστή σε αυτά τα οποία λέω. Ό,τι λέω, ό,τι λέω δημόσια σε αυτές τις χώρες, το εννοώ. Και τα ίδια πράγματα λέω και κλεισμένα των θυρών και τα ίδια λέω και δημόσια. Είμαι προσιλωμένη στη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες και αυτό περιλαμβάνει και την Αίγυπτο. Το γεγονός ότι δεν ανέφερα τα συνηθισμένα πράγματα που λέμε δεν σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι προσιλωμένη προς τα θέματα αυτά. Κυρία Λόχμπιλντερ για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των προσφύγων από την κλιματική αλλαγή. Δεν έχει προκύψει, από ό,τι ξέρω, έχετε δίκιο, καμιά συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η μία συζήτηση που νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, είναι όταν μιλάμε για τις χώρες που πλήττονται από πλημμύρες, από ε, πείνα, από δραματική αλλαγή και θυμάμαι τις δραματικές πλημμύρες στο Πακιστάν πριν από δύο χρόνια. Όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες για τα χωριά της πλημμύρας είχε γίνει πολύ σαφές ότι η κλιματική αλλαγή είχε κάποιες επιρροές στον τρόπο με τον οποίο έρχονται κάθε χρόνο οι μουσώνες και οι βροχές στα χωριά. Δηλαδή μέρη που παραδοσιακά μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την, ε, τις καιρικέ συνθήκες, δηλαδή τα μέρη που παλιά μπορούσαν να είναι βιώσιμα τα χωριά και να μην έχουν πρόβλημα, γίνονται τώρα όλο λιγότερα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνέπεια ότι μετακινούνται οι πληθυσμοί και η κίνηση των πληθυσμών είναι μία από τις απαντήσεις που γίνονται λόγω κλιματικής αλλαγής γιατί σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη πια ή να έχουν χωριά που να αντέχουν στις πλημμύρες. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο εμπίπτει στις διμερείς μας επαφές με χώρες ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, αλλά δεν έχει υπάρξει μια πλήρη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Εγώ θέλω να γίνει αυτή η συζήτηση. Και σας υποστηρίζω. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη δεν υπήρξε ποτέ μια συζήτηση ή μια κοινή θέση στο Σύμβουλο για τα θέματα αυτά. Θα το ελέγξω, αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για τα θέματα αυτά. Για συζητήσεις όπως ε, σε θέματα για το Πακιστάν, αυτά τα θέματα τα αναφέρουμε πάντα. Το Πακιστάν έχει μια στεναρή άποψη για τα θέματα αυτά και το καταγράφει αυτό κάθε φορά που συζητάμε μαζί τους αλλά μέχρι στιγμή δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Και, για το θέμα της ε, Κυρίλοφ, για το θέμα της ε, ε, εταιρικής σχέσης με χώρες της Ανατολής. Για το Ναγκόνο Καραμπάχ έχουμε ένα ειδικό εκπρόσωπο ο οποίος δαπανά πολύ χρόνο για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά στην Γεωργία ιδίω και στο Ναγκόνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτσάν το επίπεδο των επαφών μας ανεβαίνει και κατεβαίνει, ποικίλει πάρα πολύ. Εμείς ε, ανησυχήσαμε πάρα πολύ για τους νέους φράκτες που δημιούργησε η Γεωργία και το θέμα αυτό το σύντησα και με την ε, Γεωργία και με την ε, Ρωσία. Επίσης τα θέματα του Ναγκόρο Καραμπάχ προσπαθούμε πάντα να μειώσουμε τις εντάσεις και να παίξουμε ένα επικοδομητικό ρόλο για την εξέβρεση μιας μόνιμης λύσης. Ξέρουμε όλοι τι μορφή πρέπει να έχει αυτή η λύση και στην υπερνηστερία. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει επαρκή σταθερότητα στη Μολδαβία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Πραγματικά είναι σημαντικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές. Κύριε Κούκαν, σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας για τη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι υπάρχει μια ανάγκη να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα. Έκανα σαφές όμως και στους δύο πρωθυπουργού ότι θα συνεχίσουμε το διάλογο και ζητήσανε και αυτοί να συνεχιστεί ο διάλογος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή. Παραμένουν κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είναι στα Τύρανα και από αυτά που είδαμε ο Έντι Ράμα φαίνεται ότι έχει επικρατήσει και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί του όπως κάναμε και στο παρελθόν με την προηγούμενη κυβέρνηση είναι μια νέα ευκαιρία λοιπόν. Κυρία Λουξέβερ, ρωτήσατε για την Τουρκία. Νομίζω ότι απήντησα στο προηγούμενο ερώτημα για την Τουρκία. Ξέρετε με ποιο τρόπο θέλω να προχωρήσουμε. Για τη στρατηγική της ε, Μαύρης Θάλασσας επίκειται μια συνδιάσκεψη για τη Μαύρη Θάλασσα. Εγώ θα είμαι παρού, δεν θα είμαι παρούσα, αλλά θα υπάρξει εκπροσώπηση. Εμεί τονίζουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι ενεργειακοί πόροι στην περιοχή αυτή και σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Νομίζω ότι είναι, ήταν πολύ σημαντική. Προφανώς ο διάλογος θα πρέπει να προχωρήσει. Σας εύχομαι Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας το υπόλοιπο της εβδομάδας. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε κυρία Άστον. So.